Chers collègues, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. Je voudrais souhaiter Συνάδελφοι, καλώ ορίζω τον Επίτροπο Έτιγκερ. Καθίστε παρακαλώ. Μας κάνει την τιμή να έρθει εδώ, ενώπιον της Επιτροπής Προπολογισμών, για να μας παρουσιάσει τις βασικές γραμμές του σχεδίου προπολογισμού του 2018. Σχέδιο προπολογισμού που το Σώμα των Επιτρόπων μόλις υιοθέτησε. Ξέρω ότι υπάρχει φοβερή πίεση χρόνου σήμερα το πρωί, γι' αυτό θα δώσω πάρα αυτό το λόγο στον Επίτροπο, γιατί θα πρέπει μετά την ανταλλαγή απόψεων να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα στις 12 και να τα έχει στη διάθεσή του Επίτροπος, ούτως ώστε να μπορέσει να απαντήσει στις ερωτήσεις κάποιων δημοσιογράφων για μία συνέντευξη τύπου που έχει προγραμματιστεί για τις 12 και 4. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά, Επίτροπε, που είσαστε εδώ και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να παρευρεθώ σήμερα αμέσως μετά την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού στην Επιτροπή. Θα μπορέσω να σας παρουσιάσω εδώ τα βασικά στοιχεία σε εσά που είστε η αρμόδια Επιτροπή. Το σχέδιο της Επιτροπής βασίζεται σε μια ενδελεχή ανάλυση και λαμβάνει υπόψη πλήρως αυτά τα οποία εσείς και το Συμβούλιο διατυπώσατε στις προτεραιότητές σας βάσει του τριμερούς διαλόγου που έγινε τον Μάρτιο. Ο προϋπολογισμός του 2018 δεν αποτελεί καμία επανάσταση, αλλά σε μεγάλο βαθμό καλύπτει την βασική δομή και τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού όπως και το 2017. Είναι ίσως ο τελευταίος προϋπολογισμός που ε, καλύπτει πλήρως την, την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, διότι υποθέτουμε ότι οι Βρετανοί φίλοι μας ε, θα θεωρούν ε, κοινή υποχρέωση των, της πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά υπάρχουν οι άμεσες και έμεσες συνέπειες της εξόδου των Βρετανών φίλων μα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με όλε τι συνέπειε και για τον προπολογισμό. Κατά τι τελευταίε εβδομάδε είδαμε πόσο εντατικά γίνονται ε, οι συζητήσεις για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση είναι δική σας επιτυχία κατόπιν ετοιμάτων ε, του Κοινοβουλίου από το 2013, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν το επιθυμούσε το Συμβούλιο. Έγινε όμως στη συνέχεια αποδεκτή και νομίζω ότι είναι προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και προς όφελος των κρατών μελών γιατί η ενδιάμεση αναθεώρηση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, ιδιαίτερα χρήσιμο στο Συμβούλιο έγινε αποδεκτή αυτή ε, η πρόθεση και θα υπάρχουν και οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και λόγω και της εκλογικής περίοδου το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να αποδεχθεί πλήρως τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία πολιτικής και βάσει της αρχής των πιθανοτήτων για τη διαδικασία που ακολουθείται στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο εμείς παρουσιάσαμε την ενδιάμεση αναθεώρηση. Εκ παραλληλού διαμορφώσαμε για το Συμβούλιο και για το Κοινοβούλιο στοιχεία για το τι θα συμβεί εάν αποκλίνουμε από τη θεωρία των πιθανότητων την οποία έχουμε αποδεχθεί. αν δεν θα μπορούσε δηλαδή να γίνει αποδεκτό αυτό το σχέδιο προπολογισμού βάσει τη ενδιάμεση αναθεώρηση, τι είδου ε, αλλαγέ ε, θα επέλθουν. Και τι τροποποιήσεις θα επέλθουν χωρίς ενδιάμεση αναθεώρηση στο σχέδιο της Επιτροπής τι σημασία έχουν όλα αυτά και τι επιπτώσεις θα έχουν για τις δαπάνες και για τα κοινοτικά προγράμματα. Τους υπολογισμούς μας όμως τους κάνουμε με την υπόθεση ότι θα έχουμε ένα εγκεκριμένο σχέδιο ενδιάμεσης αναθεώρησης μετά τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο. Έχουμε ορισμένες προτεραιότητες ένας τομέας δαπανών που αφορά την μετανάστευση και τους πρόσφυγες που δίνει έλεγχο στα σύνορα και προστασία στα σύνορα για τα ε, άμεσα θυγόμενα κράτη-μέλη. Έχουμε επίσης κονδύλια για την ανάπτυξη και για την απασχόληση των νέων. Και η ενδιάμεση αναθεώρηση θα είναι μεγάλη ε, διευκόλυνση και για τους δύο αυτούς τομείς, διότι παρέχει ευελιξία, μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι πριν, με, μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ των ετών του προϋπολογισμού και μεταξύ ε, των ε, τομέων του προϋπολογισμού μέσα σε κάθε έτος. Στα προτινόμενα μέτρα για τις υποχρεώσεις, Έχουμε 160,6 δισεκατομμύρια αύξηση σε σχέση με το 2017 αύξηση της τάξης του 1,4%. Ο προϋπολογισμός φτάνει ε, σε ένα επίπεδο που δεν είχε φτάσει, όπου δεν είχε φτάσει μέχρι τώρα. Υπάρχει και περιθώριο ελιγμών για τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και για νέες ανάγκες που δεν έχουν προκύψει μέχρι τώρα. Τα προτινόμενα κονδύλια για τις πιστώσεις πληρωμών είναι 145,4 δισεκατομμύρια και αυτό σε σχέση με, τον, με το τρέχον έτος, το 2017, σημαίνει αύξηση 8,1%. Φαίνεται μεγάλη αυτή η αύξηση. σας θεωρώ εταίρους για μια δίκαιη ε, διαπραγμάτευση. Αυτό το 8,1% για το 2018 σε σχέση με το 2017 σημαίνει υψηλότερες πιστώσεις πληρωμών και αυτό έχει σχέση με την ταχύτητα διεξαγωγής του επταετούς ε, πλαισίου. κάποια ε, ε, κονδύλια ε, που εγκρίθηκαν αργά το 2013, το Δεκέμβριο του 2013, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν το 2014. Δεν είχε ξεκινήσει η πραγματική πορεία εφαρμογής. Τώρα όμως βρισκόμαστε απολύτως σε πορεία λειτουργική, πάντοτε στα πλαίσια του ανωτάτου ορίου, πάντοτε στα πλαίσια του πλαισίου που έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο, αλλά έχουμε ανακτήσει την πλήρη ταχύτητά μας, επομένως μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουν προγραμματιστεί για την επταετή περίοδο. Το 8,1% εκφράζει ότι τα έργα τα οποία έχουμε αποφασίσει θέλουμε να τα υλοποιήσουμε, θέλουμε ε, να τα υλοποιήσουμε προς όφελος της αγοράς εργασίας και της ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος της ανάπτυξης ε, κατά της στασιμότητας με σχετικά καλές προοπτικές ανάπτυξης για το 2018, ε, την οποία και θέλουμε να βελτιώσουμε. Επαναλαμβάνω, το 8,1% δεν είναι ε, μια ε, άποψη της Επιτροπής που ξαφνικά θέλησε να δώσει μια τεράστια ανάπτυξη. Είναι κάτι που βρίσκεται εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Και τα κονδύλια αυτά θα αφορούν μόνο προγράμματα τα οποία ε, συμπεριλαμβάνονται στο επταετές πλαίσιο. Έχουμε κάποιες προτεραιότητες για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2018 για να λάβουμε υπόψη μας γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως σας είπα στην αρχή, θέματα μετανάστευσης, μεταναστευτικές ε, ροές, θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας, αστάθεια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε γειτονικέ ε, περιφέρειες. Δεύτερον, στρατηγικές επενδύσεις, έρευνα, καινοτομία, ανάπτυξη, απασχόληση, ιδίως για τους νέους. Για το πρώτο που ανέφερα, ασφάλεια και μετανάστευση. Το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ευρωπαϊκή απόκριση στη μετανάστευση και την κατάσταση ασφάλειας και στο εσωτερικό και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έξω από τα σύνορα των 28 κρατών μελών μας. Για την περίοδο 2015 έως το 2018 το συνολικό ποσό αυξάνεται κατά 22, φτάνει στα 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Γρήγορα προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε σε νέες ανάγκες και σε νέες προκλήσεις και υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη τα οποία πλήττονται περισσότερο πράγμα το οποίο αποτελεί και ένδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα ενδυναμώνονται, ενισχύονται και ε, τους χορηγούμε τα απαραίτητα οικονομικά μέσα και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας για το συντονισμό ε, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας δίδονται επίσης τα κατάλληλα ε, κονδύλια. Επίσης, μέσα λαμβάνονται και για την αντιμετώπιση της, ε, των αιτιών της μετανάστευσης σε τρίτες χώρες για να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές και για να βοηθήσουμε τις χώρες ε, που πλήττονται περισσότερο από όλες. Όσον αφορά την ασφάλεια, έχουμε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τα ευρωπαϊκά σύνορα και τις ευρωπαϊκές ακτές, το σχέδιο προϋπολογισμού λαμβάνει υπόψη διάφορα στοιχεία. Ένα κοινό σύστημα ασύλου και την επεξεργασία του κοινού συστήματος ασύλου, καλύτερη διαχείριση των συνόρων, δημιουργία ενός συστήματος ενημέρωσης και πληροφόρησης για θέματα ε, ταξιδίων, ε, μετακινήσεων, ε, θεωρήσεων διαβατηρίου κλπ. Ούτως ώστε να έχουμε τους κατάλληλους ελέγχους και τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Λαμβάνοντας υπόψη και την κατεύθυνση που θέλουμε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασύλου να γίνει ένας πραγματικός οργανισμός ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα καλύπτει όλες τις απαιτήσει. Έχουμε 200 εκατομμύρια για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν ε, ε, τρεις τομείς που ξεπερνάνε το όριο κατά 0,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτοί είναι τομείς όπου χρησιμοποιούμε μέσα ευελιξίας, τα οποία είναι απαραίτητα. Μέσω της ενδιάμεσης αναθεώρησης, αυτή η ενίσχυση με τα σχετικά κονδύλια καθίσταται δυνατή. Στον τομέα 4 προτείνουμε 1,9 δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση των αιτιών της μετανάστευσης, ανθρωπιστική βοήθεια, βοήθεια σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών κλπ. Είναι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και ίσως προκύψουν και νέες ανάγκες, ίσως να υπάρξουν εκ νέου μεγάλες ε, προσφυγικές ροές. Και γι' αυτό στον τομέα η Ευρώπη στον κόσμο έχουμε 230 εκατομμύρια τα οποία θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε σε μελλοντικέ ανάγκες για να είμαστε ε, ε, αξιόπιστη εταίροι έναντι και των γειτόνων μας, όπως είναι και η Τουρκία. Ξέρετε ότι υπάρχει μια συμφωνία τριών δισεκατομμυρίων. Τα χρήματα αυτά δεν δίδονται σε παλάτια που χτίζονται στην Άγκυρα, αλλά δίνονται για καλύβες, για σκηνές όπου ζουν ε, πρόσφυγες για να αντιμετωπίσουν ε, προβλήματα που αντιμετωπίζουν για τη διατροφή τους, για τη διαμονή τους, για καθαρό νερό, για διατροφή. Αυτά τα τρία δισεκατομμύρια θα εξαντληθούν πριν από το τέλος του έτους. Εάν υπάρξει μια νέα συμφωνία προς όφελος των προσφύγων που βρίσκονται σε στρατόπεδα στην Τουρκία, και αν ε, οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται βοήθεια, ανεξάρτητα από τη στάση μας έναντι της, της κυβέρνησης ε, στην Άγκυρα, ίσως θα πρέπει να δώσουμε κάποια επιπλέον χρήματα για να δείξουμε την διάθεσή μας ε, για σωστές διαπραγματεύσεις. θα πρέπει να προσθεθούν κονδύλια, ούτω ώστε να υπάρξει μια παράταση της συμφωνίας με τα επιπλέον 3 δισεκατομμύρια που θα απαιτούσε μια νέα συμφωνία. Βιώσιμες επενδύσεις και νέα γενεά είναι η άλλη προτεραιότητα. Στον τομέα 1 Έχουμε κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την επάνωδο της ανάπτυξης. Εδώ το 48% του συνολικού πλαισίου ε, το έχουμε συμπεριλάβει εδώ για πολλά προγράμματα τα οποία είναι σημαντικά για όλους μας. Για το Horizon 2020, για το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας. Αύξηση 770 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό γίνεται διότι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για σας αυτό το πρόγραμμα και πόσο σημαντικό είναι για την κοινότητα των ερευνητών στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα Horizon 2020 ε, είναι ευρύτατα αποδεκτό από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για την υλοποίηση του σχεδίου Juncker είναι απαραίτητες αυτές οι επενδύσεις. Και γι' αυτό και αναδρομικά μπορούν να δοθούν κάποια κονδύλια. Για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, το Connecting Europe Facility, προσθέτουμε 220 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό με την πρότασή μας και για το Erasmus Plus δίνουμε 200 εκατομμύρια επιπλέον. Για το FC για την, ε, το τελευταίο κομμάτι ε, ε, του FC2 και για την παράταση του FC2 προστίθενται χρήματα στον προϋπολογισμό και για το Wi-Fi for Europe ώστε να υπάρχουν πολύ περισσότερα σημεία Wi-Fi και προσθέτονται στο σχέδιο προϋπολογισμού τα αντίστοιχα ε, ποσά. Το θέμα της έρευνας στον τομέα της άμυνας είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία στον τομέα της άμυνας μέσω του συντονισμού, μέσω μείωσης ε, των διαφορετικών ειδών ε, οπλισμού στα επόμενα τρία χρόνια, το 2018, 2019 και 2020, έχουμε βάλει στον προπολογισμό 90 εκατομμύρια, εκ των οποίων 40 μέσα στον επόμενο χρόνο. Αυτά θα είναι προπαρασκευαστικά μέτρα για την έρευνα στον τομέα της ε, άμυνας. Στον τομέα της έρευνας δεν έχουμε πρόβλημα με τις αρμοδιότητες βάσει της συνθήκης. Στην ε, άμυνα έχουμε περιορισμούς, αλλά στην έρευνα για την άμυνα δεν έχουμε περιορισμούς. Στο Horizon 2020 έχουμε για μη στρατιωτικούς σκοπούς έρευνα. Εδώ έχουμε ένα επιπλέον ποσό έρευνα για την έρευνα για πιλωτικά έργα για τον τομέα της ε, άμυνας. Ενημέρωσα και τους ε, συναδέλφους σας στην Επιτροπή Πολιτισμού σε μια συνάντηση σε σχέση με αυτό το οποίο προτείνεται για, την Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει ευκαιρίες για νέους οι οποίοι θα προσφέρουν εθελοντική εργασία και για τα τρία χρόνια μέχρι ε, το τέλος της επέτους περίοδου έχουμε 342 εκατομμύρια. 89 εκατομμύρια μέσα στον επόμενο χρόνο, το 2018 και μέσω ανακατατάξεων και μέσω νέων κονδυλίων προτείνεται αυτό το ποσό για τα επόμενα χρόνια. Θα μπορούσα να σας παραθέσω πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Έβαλα μόνο την πρωτοβουλία απασχόλησης για τους νέους, αυξάνονται τα κονδύλια τα οποία ανέμενε και το Κοινοβούλιο. ...1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ε, είναι το συνολικό ποσό και παίζει η πρωτοβουλία αυτή πολύ σημαντικό ρόλο. Περνάω τώρα στις βιώσιμες επενδύσεις σα είπα ότι για τα μέσα πληρωμών, για τι υποχρεώσει πληρωμών, ε, είχαμε μια αύξηση 8,1%. Μια καλή είδηση είναι ότι τα τελευταία χρόνια ε, έχουμε επεξεργαστεί όλα τα κονδύλια τα οποία δεν είχαν πληρωθεί και έχει ε, μειωθεί το ποσό των ε, ε, δαπανών προς ε, πληρωμή. Και εσείς το επιδιώξατε αυτό. Και τώρα πλέον ο προϋπολογισμός μας βρίσκεται στην ταχύτητα πορείας την οποία απαιτούν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτή την αυξημένη ταχύτητα λοιπόν έχουμε αυξήσει τα κονδύλια τα οποία δίδονται κατά 26 περίπου της 100. Αυτά είναι πληρωμές ε, για επενδύσεις, για διαθροτικές επενδύσεις. Και αυτό συμπεριλαμβάνεται στην αύξηση του 8,1% που σας ανέφερα προηγουμένως. Αυτά τα οποία διεξήχθησαν κατά το 2014-2015 δεν θα επαναληφθούν κατά τα επόμενα χρόνια. θα ακολουθήσουν οι πληρωμές οι οποίες ε, απαιτούνται ούτω ώστε από τώρα μέχρι το τέλος ε, του δημοσιονομικού πλαισίου να καταβληθούν αυτά τα οποία οφείλονται και να μην υπάρξει καθυστέρηση πληρωμών. Περνώ τώρα σε διοικητικές δαπάνες. Είχαμε μία μείωση του προσωπικού κατά 5% που ήταν πακέτο της δέσμης μέτρων για τον προϋπολογισμό από το 2013 μέχρι το 2017 και τα περισσότερα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εφαρμόσει τη μείωση αυτή. Είχαμε μία μείωση 1.947 θέσεων, εκ των οποίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωση 1.254 θέσεων, η Επιτροπή που έχει, είχε τη, τη μεγαλύτερη μείωση θέσεων. Για τους διάφορους οργανισμούς που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η δέσμευση μείωσης θα έχει καλυφθεί μέχρι το τέλος του 2019. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Κοινοβούλιο θα δείξουν τα στοιχεία αυτά μέσα στον επόμενο χρόνο. Συνεχίζουμε με την πορεία εξοικονόμησης δαπανών. Υπάρχουν όμως δαπάνες οι οποίες είναι απαραίτητες για υποδομή πληροφορικής, παραδείγματο χάρη, κάτι το οποίο αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Θέλουμε να μπορούμε να υπεραμεινθούμε των εγκαταστάσεών μας έναντι κυβερνοεπιθέσεων. Ξέρουμε ότι τα κτίρια μας και οι εγκαταστάσεις μας τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Ε, θέλουμε να έχουν καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Και αυτό θα το επιτύχουμε με ε, ορισμένα, ορισμένες ανακαινήσεις σε κάποιες περιπτώσεις για βελτίωση των λειτουργικών δαπανών. Επίσης θα λυθούν υπόψη ε, τα θέματα των συντάξεων και βέβαια δεν μιλάμε για μειώσει σε αυτόν τον τομέα γιατί όλοι οι συνεργάτες μας και όλοι οι υπάλληλοι έχουν ε, δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια ώστε να ε, δικαιούνται την δίκαιη αμοιβή τους. Πληρώνουμε τους επαλλήλους μας κατά την ενεργό επαγγελματική τους ζωή με ε, την αμοιβή τους και επειδή είχαμε ε, μια γραμμική αύξηση ε, του προσωπικού είχαμε μια δυναμική γραμμική αύξηση του προσωπικού και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μεγαλύτερη κλίμακα, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Άρα θα έχουμε και μια, ένα νοδικό κύμα στις συντάξεις. Στον προπολογισμό του 2018 έχουμε αύξηση 3,1%. Είναι ποσοστά που θα συνεχίσουμε να βλέπουμε να αυξάνονται κατά τα επόμενα χρόνια, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το ανωδικό κύμα στις συντάξει. Και αυτό θα αποτελεί στρατηγική στον προϋπολογισμό που θα ακολουθήσουμε κατά τις συζητήσεις για τα επόμενα πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια. Θα ήθελα να πω ακόμη δύο λόγια για την έννοια του προϋπολογισμού που είναι προσανατολισμένος στα αποτελέσματα. Προσπαθούμε να έχουμε όλο και καλύτερη υποβολή εκθέσεων. με εκθέσεις και ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού, τα οποία προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε μία σύνοψη αυτών τα οποία ήδη σας παρουσίασα. Βλέπετε εδώ τους διάφορους τομείς. Βλέπετε τις πιστώσεις υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών. Και βλέπετε και τα μέσα ευελιξίας πώς μας βοηθούν να καλύψουμε νέους τομείς δαπανών. Τέλος, με την ε, πρόταση αυτή πιστεύω ότι ε, βελτιώνουμε τις προοπτικές. Ελπίζω ότι θα δεχθείτε αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού. Δεν, θα, δεν φαντάζομαι ότι θα τα δεχτείτε 100% αλλά νομίζω ότι θα, θεωρείτε, θα θεωρήσετε ένα ε, βάσιμο και αξιόπιστο σχέδιο προϋπολογισμού αυτό που σας παρουσίασα. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους και τους συζητητές και όλες τις πολιτικές ομάδες ε, κατά τις επόμενες εβδομάδες να ε, συμμετάσχετε σε έναν ε, επικοδομητικό διάλογο, ούτως ώστε να τηρήσουμε τις προθεσμίες, να εγκριθεί ο προϋπολογισμός μας εγκαίρος, γιατί αυτό το αποκλίνεται στις προσδοκίες των πολιτών μας, για να δείξουμε ότι όντως προσθέτουμε προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Merci, monsieur le Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την παρουσίαση πολύ συνοπτική, απόλυτα ξεκάθαρη, που φαντάζομαι θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους, στους Ευρωπαίους πολίτες να καταλάβουν τι είναι ο προϋπολογισμός και σε ποιους στόχους ανταποκρίνεται. Πολύ ωραία. Θα πρέπει να σεβαστούμε το χρόνο Για να κλείσουμε θα σας δώσουμε το λόγο στις 12 ε, ή 12 και 5. Γι' αυτό λοιπόν οι ομιλητέ θα πρέπει να είναι πολύ λακωνικοί. Ξέρω ότι οι ασκήσεις ε, ελέγχου του προπολογισμού ε, είναι κατάλληλες για να ασκήσουμε όλη η αυτοπιθαρχία. Τρία λεπτά λοιπόν έχουν οι εισηγητέ και ενάμιση ισχυώδει εισηγητέ. Ο κ. Μουρεσάν, ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε, Πίτρο Πέτιγκερ, στο Κοινοβούλιο και σε ευχαριστώ που παρουσιάσατε το σχέδιο προπολογισμού. Από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε από τα όσα μας είπατε, το σχέδιο προϋπολογισμού που μας παρουσιάζεται έχει τις βασικές προτεραιότητες που ζήτησε το Κοινοβούλιο στις κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετήσαμε το Μάρτιο. Έχουμε δύο βασικές προτεραιότητες για το προϋπολογισμό του 2018. Πρώτον, ε, ανάπτυξη και θέση απασχόλησης. Δεύτερον, ασφάλεια των πολιτών γιατί αυτό πιστεύουμε ότι οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουν, ε, θέλουν. Να χρησιμοποιήσουμε του ελάχιστου πόρου που έχουμε για αυτά τα θέματα. Επίση, έχετε ένα προλογισμό ο οποίος ε, καλύπτει τι νέε ανάγκε λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων. Υπάρχουν, λοιπόν, υπάρχει προσοχή στην άμεση γειτονία μα και στον προπολογισμό και είναι σωστό αυτό. Και εμεί στο Κοινοβούλιο πάντα είχαμε τη θέση ότι οι νέες προτεραιότητε, οι νέε προκλήσεις που δεν είχαμε προβλέψει το 2013, όταν αποφασίστηκε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να καλυφθούν με νέα κονδύλια. Γι' αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω την εισαγωγή από την Κομισιόν της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και αυτό μπαίνει ήδη στο σχέδιο προπολογισμού. Αυτό ήταν συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και τώρα πιστεύουμε ότι και το Συμβούλιο και περιμένουμε και το Συμβούλιο να κάνει, να κάνει αυτά που πρέπει. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο μα είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γραφειοκρατική και παίρνει αργά τι αποφάσει τη. Ε, ελπίζουμε λοιπόν να μην μπλοκάρει ε, τα πράγματα στο Συμβούλιο το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτή τη σημαντική αναθεώρηση, ούτω ώστε να έχουμε περισσότερου πόρου για, για το μηχανισμό διευκόλυνση τη Ευρώπη, το ορίζοντα 2020, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή που ενδυναμώνουν την οικονομία μα. Τώρα, σύντομα για τον προπολογισμό για τον τομέα 1. Όπως σας είπα, η ε, ανάπτυξη και η θέση απασχόλησης θα πρέπει να είναι ένας, μία από τις προτεραιότητες του προπολογισμού του 2018. Ε, μας ενθαρρύνουν οι αυξήσεις που μας προτείνεται στον ορίζοντα 2020, στον Erasmus, για το Erasmus ειδικά. Πάντα έχω πει ότι η επένδυση στο Erasmus ε, καθιστά την εργατική μας δύναμη πιο ανταγωνιστική, πιο ικανή να μετακινείται ε, και μας αρέσει και η αύξηση στο Connecting Europe Facility. Θα μας πείτε περισσότερα για τις ε, μειώσεις του 2,9% στο κόσμο που προτείνεται. Είναι συνέπεια της αύξησης ε, του προϋπολογισμού του περσινού ε, στον τομέα 1β, η αύξηση των πληρωμών, 25%. Να μας πείτε περισσότερα για το αν πιστεύετε ότι Αρκούν αυτά για να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες, δεδομένου του ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα θα τρέχουν ε, πλήρως ε, το 2018, θα έχουν φτάσει σε ε, ταχύτητα πορείας. Επίσης θα πρέπει να εγκριθούν οι διαχειριστικές αρχές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνει η Κομισιόν για τα ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα, να φτάσουν στο επίπεδο που πρέπει και τα λεφτά να συνεχίσουν να ρέουν. Στο τομέα 2, ε, καλωσορίζω τις αυξήσεις στα προγράμματα που προτείνεται. Επίσης, το επιπλέον περιθώριο των 730 εκατομμύριων ευρώ που προτείνεται θεωρείται ότι είναι αρκετά για να ανταποκριθούν στα πρόβλεπτα στον τομέα της γεωργίας, όπως παραδείγματος χάρη η κρίση των γαλακτοκομικών που αντιμετωπίσαμε πέρυσι, θα πρέπει να είμαι στο πλευρό των ε, γεωργών εάν ε, τους χτυπήσει κάποια κρίση. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, για τον τομέα ναι, η αύξηση στις, ε, στους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν ευθύνε στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών, ε, όπως ζήτησα και εγώ στις ε, προσανατολισμούς μου, εσείς προτείνετε ε, για το ΕΑΣΟ, το Europol και το EU Lisa σημαντικές αυξήσεις, και εγώ το ήθελα, σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα για τη μείωση όμως που προτείνετε για τα προγράμματα AMIF, ISF. Θεωρούμε ότι τα λεφτά είναι κατάλληλα, είναι ρεαλιστικά, καλό θα ήταν να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου τελείωσε η κρίση ε, των προσφύγων και μπορούμε να ενισχύσουμε πλέον τα σύνορά μας και να εμποδίσουμε την επόμενη κρίση ε, επενδύοντας περισσότερο. Αλλά ας μην είμαστε υπεραισιόδοξοι. Μας αρέσουν και τα 40 εκατομμύρια που προβλέπετε για τις προπαρασκευαστικές δράσεις για την άμυνα. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ε, ξοδεύουμε λεφτά μία φορά, όχι 28 φορές ε, το κάθε κράτος μέλος χωριστά και να μοιραζόμαστε τα αποτελέσματα όπως είναι σωστό μεταξύ εταίρων. Αυτά, Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ. Από ό,τι μπορώ να κρίνω, το σχέδιο προπολογισμού ευθυγραμμίζεται με τις βασικές προτεραιότητες που ζήτησε το Κοινοβούλιο, αλλά σαφώς υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου θα θέλαμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες ε, τις επόμενες εβδομάδε και περιμένω τις ε, συζητήσεις και την αλληλεπίδραση με την Κομισιόν και ίσως θα χρειαστούν να γίνουν και κάποιες προσαρμογές στον προϋπολογισμό. Ε, ίσως για να τα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο θα πρέπει να κάνουμε κάποιους, κάποιες αλλαγές. Ελπίζω όμως να συμφωνήσουμε με τον Συμβούλιο. Ευχαριστώ για την, για το, την προσπάθεια λακωνικής παρουσίασης. Ε, στο, αυτό ήταν ο γενικός εισηγητής, η κυρία Ντανιέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε που, για αυτή την παρουσίαση. Ο Γενικός Εισηγητής ε, κάλυψε πολλές από τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο πολύ θετικό στοιχείο, το ότι η Κομισιόν θέλησε να βάλει στο σχέδιο προπολογισμού την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Ξέρουμε ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα από το Συμβούλιο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα και θεωρώ ότι κανονικά θα μας διευκολύνει τη ζωή. Οι προτεραιότητες που, βάλουμε, που βάλαμε αντικατοπτρίζονται παραδείγματος χάρη επενδύσεις, ε, απασχόληση των νέων, εράσμους, ε, μετανάστευση, ε, χρησιμοποιούνται αρκετά από τα περιθώρια. Ε, μένει ένα δισεκατομμύριο περιθώριο για τους, για τους τομείς 2 και 4 χωρίς εκτέλεση. Υπάρχει μια αύξηση των πληρωμών. Ελπίζουμε τώρα να μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια και να μην επιστρέψουμε λεφτά στα κράτη-μέλη όπως κάναμε τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να δούμε το σχέδιο του προϋπολογισμού με περισσότερη προσοχή. Να σας κάνω όμως ήδη κάποιες ερωτήσεις. Στο σχέδιο για την αναθεώρηση του πολιτού του δημοσιονομικού πλαισίου υπάρχουν αύξηση σε κάποιες προτεραιότητες. Όντως. Όμως υπάρχουν και κάποιες ε, ανακατατάξεις σε ποιε κατηγορίες, σε ποια προγράμματα θέλω να μου πείτε, πήρατε από ποια προγράμματα μάλλον πήρατε προγράμματα για να τα πάτε στην ορίζοντα 2020 ή για να τα πάτε στο Έρασμους. Έχετε μπροστά σα τα νούμερα για την χρήση ε, του μηχανισμού ευελιξίας Και όταν ε, εγκριθεί η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου μπορούμε να κάνουμε επίσης κάποιες μεταφορές. Και με ποια εργαλεία το Κοινοβούλιο μπορεί να ενισχύσει τα προγράμματα που κατά την άποψή του είναι προγράμματα προτεραιότητας που είναι πιο σημαντικά. Αυτά ευχαριστώ. Ο κ. Κολμέλη έχει το λόγο τώρα. λάμβανε τον λόγο ο συζητητής για τα άλλους τομείς, τα άλλα τμήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, βεβαίως. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τον Επίτροπο. Αναγνωρίζω ότι έχει πάρα πολλούς περιορισμούς από τον πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά βλέπουμε το 1% αύξηση στις πληρωμές και θα θέλαμε να δούμε λεπτομερώς ε, τι, ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Αλλά δύο γενικά σχόλια θα ήθελα, κύριε Επίτροπε, να σας πω. Θέλω να σας ε, συγχαρώ, διότι κρατήσατε στο πρόγραμμα εγκαίρως το θέμα των ανεξόφλητων λογαριασμών. Ελπίζω να μπορέσετε εν καιρό ε, να το λύσετε το θέμα αυτό και θα σας συγχα... συγχαρώ τότε. Βεβαίως εγκρίνω αυτό την εντύπωση που έχετε ε, για την ε, αντίληψη της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Θα πρέπει ό,τι ξοδεύουμε να προσθέτει ευρωπαϊκή αξία και με τις προτεραιότητες ε, βεβαίως είμαι ικανοποιημένο και νομίζω ότι αυτό θα το επιτύχετε. Σχετικά με την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα έχω τρία σημεία. Πρώτον, ε, τις λεπτομέρειες όσον αφορά ε, το FC2, το FC1 ήταν ικανοποιητικό, θα ήθελα τις λεπτομέρειες ε, για αυτό το Ταμείο 2. Επίσης θα ήθελα περισσότερες αναφορές σε αυτό που ονομάζω ανάπτυξη πράσινη και ευφυή, έξυπνη ανάπτυξη, ε, όσον αφορά ε, την ανεργία, δεν ε, διαφωνούμε με τις απόψεις σας, αλλά θέλουμε ορισμένα προγράμματα στα κράτη-μέλη απασχόλησης και νομίζω ότι τα προγράμματα αυτά δεν δίνουν αποτελέσματα που είναι προστιθέμενη αξία. Ένας νέος που θέλει εκπαίδευση, κατάρτιση και θέλει μια αναπτυσσόμενη οικονομία που να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Βλέπω ότι ανταποκρίνεστε στις ανησυχίες του κοινού για τα θέματα μετανάστευσης, ασφαλείας, με δαπάνες βεβαίως θα πρέπει αποτελεσματικά να είναι τα αποτελέσματα. Ως προς τη δίκηση σας συγχαίρω ε, για την ε, μείωση προσωπικού που προβλέπετε αλλά βεβαίως χρειαζόμαστε ε, να ικανοποιηθούν περισσότερες ανάγκες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και νομίζω ότι το πήρατε το μήνυμα βεβαίως ε, ως προς τις συντάξεις. Ε, έχουμε ένα θέμα που πρέπει να ερευνηθεί ως προς τα άλλα τμήματα, τους άλλους τομείς του προϋπολογισμού. Θα δούμε και τους επόμενους μήνες τι θα, τη συνέχεια και θα μπορέσουμε ίσως τότε να έχουμε και άλλα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μικρόφωνο, μικρόφωνο παρακαλώ. Νο, όχι. Εάν ήταν παρούσα, νομίζω ότι θα είχε επιμείνει για τις πληρωμές, κύριε Επίτροπε, διότι χθες είχαμε μια συνεδρίαση με τον Γιάνν Σκελέρ, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα διορθωτικού προϋπολογισμού 2 ε, για το 2017 που έδειξε το 2016 σε σχέση με τις προβλέψεις οι, μειώ... πληρωμές μειώθηκαν κατά 12 δισεκατομμύρια που είναι σημαντικό ποσό. Αύριο λόγω της επίπτωσης γιογιό θα έχουμε ένα άλμα ε, στις, ε, στις αιτήσει πληρωμών ή μήπως υπάρχει έλλειψη όρεξης από τους ε, διάφορους πρωταγωνισμούς οι οποίοι έχουν περιορισμούς δημοσιονομικούς και ξέρουν ότι η βοήθεια ευρωπαϊκή είναι μέρος της χρηματοδότησης και ότι να δεχθούμε τη βοήθεια την ευρωπαϊκή είναι σαν να έχουμε πρόσθετες δαπάνες. Θέλουμε λοιπόν διευκρινήσεις για αυτό το θέμα και ως προς την απασχόληση των νέων νομίζω ότι η κυρία Ζολμακή θα είχε αναφερθεί στα προγράμματα που ενέταξε η Επιτροπή για το 2018 και πέραν αυτού του έτους, δηλαδή να αναλάβει ένα πολιτικό πρόγραμμα για την κινητικότητα των μαθητευομένων στην Ευρώπη, πράγμα που απαιτεί ε, ε, Erasmus πλάσα, ε, δηλαδή πρόσθετα κονδύλια για το Erasmus να, να διευρυνθεί το κονδύλιο, όπως υπενθύμησε ο Γενικός Εισηγητής, ε, διότι πάρα πολλά αιτήματα που είναι επιλέξιμα, πολλές αιτήσει δεν ικανοποιούνται όπως στον τομέα της έρευνας. Χθε είχαμε μια επιτροπή παρακολούθησης ε, για το Horizon 2020. Ε, προβλέψατε 11 δισεκατομμύρια ακόμα και οι υπηρεσίες της Επιτροπής που ασχολούνται με την έρευνα περιμένουν το κονδύλι αυτό με ενδιαφέρον. Δίνω το λόγο στην κυρία Ντιριεντά ή στον κύριο Ομαρζή που δεν είναι εδώ παρόντες. Ε, δίνω λοιπόν για τους πράσινους το λόγο στην κυρία Εμρεταραγκ. Ευχαριστώ στον κύριο. Ε, κύριε Επίτροπε, θα μπορούσα να πω πολλά θετικά πράγματα για το σχέδιο προϋπολογισμού ε, για την μείωση των διοικητικών δαπανών, αλλά για να χρησιμοποιήσω παραγωγικά το χρόνο μου, έχω δύο ερωτήσεις, δύο ερωτηματικά σχετικά με τις προθέσεις σας. Πρώτα απ' όλα, πρόσφατα ήμουνα σε μια διάσκεψη ε, και ο πρόεδρος της Φινλανδίας δήλωσε ότι υπάρχουν πολύ ε, μεγαλύτερες απειλές στην ασφάλεια από την τυχοδιοκτισμό της Ρωσίας ε, και την ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Δύο χώρες δεν αναγνωρίζουν την κλιματική αλλαγή και σε αυτή τη χρονική στιγμή νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αποδώσει μεγαλύτερη σημασία στην χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το κλίμα και ξέρουμε όλη την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και βλέπουμε ε, τις Ηνωμένε Πολιτείες που δεν θέλουν ε, να ε, τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το κλίμα. Η ερώτησή μου, ε, νομίζετε ότι υπάρχει δυνατότητα για τον προϋπολογισμό του επομένου έτους να έχουμε μια χρηματοδότηση τούρμπο στον τομέα αυτό. Και δεύτερον, νομίζω, αν κατάλαβα σωστά, σε αυτό το σώμα, ε, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, τα πρόσθετα κονδύλια είναι περίπου 80% προέρχονται από το πρόγραμμα Erasmus Plus και διαρωτώ με, δεδομένου ότι το Erasmus Plus ε, θα είναι από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ακόμη δυνατότητα να, να θεωρήσουμε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ε, του σώματος αλληλεγγύης και να αφήσουμε το Εράσμους ως έχει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Οι άλλοι σκιώδεις εισηγητές δεν είναι παρόντες. Έχω εδώ έναν κατάλογο ε, Γιάν Ολμπριχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο. Βεβαίως ε, θέλουμε να έχουμε λεπτομέρειες των προτάσεών σας. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι ότι είναι προδραστικός ο Επίτροπος σχετικά με την συμπεριφορά του Συμβουλίου θα θέλαμε να χαιρετήσουμε τις αποφάσεις σας. Είναι πολύ επικίνδυνες αυτές οι αποφάσεις, αλλά το, τις λύσεις αναθεώρησης τις βάλατε μέσα στον προϋπολογισμό και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σχετικά με την δυναμική όλης της διαδικασίας, διότι χωρίς αυτό κανείς δεν θα δει τις πραγματικές επιπτώσεις της αναθεώρησης ενώ έτσι τις βλέπουμε. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο όπου μπορούμε να δούμε στον προϋπολογισμό έχετε νέα στοιχεία για το επόμενο πλαίσιο όταν έχετε τις προπαρασκευαστικές δράσεις για την ασφάλεια και την άμυνα. Αυτό έρχεται, είναι τα πρώτα βήματα και για μας είναι ένα πολύ σημάδι πολιτικό ότι αρχίζετε το 18 αλλά θα έχετε προτάσεις πιο ενισχυμένες ε, για το επόμενο πλαίσιο. Το τρίτο στοιχείο, ίσως όχι για σήμερα, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι μια νέα ιδέα, 9 εκατομμύρια, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι νέα πρωτοβουλία. Το θέμα είναι ε, τι θα είναι αυτή η πρωτοβουλία. Νομίζω ότι δεν θα είναι για ένα έτος, αλλά και για τα επόμενα έτη. Ποια είναι η όλη διαδικασία για αυτό το σώμα και τελευταία παρατήρηση ε, σχετικά με τις καθυστερήσεις ε, στις πιστώσεις πληρωμών, τις ισορευμένες καθυστερήσεις. Το 17 έχουμε χαμηλά επίπεδα και τώρα έχουμε συν 25%. Αλλά 25% από πολύ χαμηλά είναι ακόμη πάρα πολύ χαμηλό. Υπάρχει το θέμα, είναι ε, αρκετό αυτό διότι ε, τον, για το 18, 19 ή 20 αν θέλουμε, αν έχουμε ένα συν 5% πόσο περισσότερο θα έχουμε το 19, το 20 για να αποφύγουμε ε, την ε, συσσόρευση εκκρεμωτήτων, καθυστερημένων εκκρεμωτήτων. Ευχαριστώ. Ο Γιάνς Γκέιερ, ο τελευταίος ε, παρεμβαίνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις, πολλές παρατηρήσεις. Θα προσπαθήσω να περιορίσω τα σχόλιά μου. Το πρώτο για την εγγύηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το FC2. Πρέπει να κινητοποιήσουμε 8 δισεκατομμύρια για να μπορέσουμε να επιτύχουμε 16 δισεκατομμύρια. Αν θέλουμε να το επιτύχουμε αυτό μέχρι το 2020, θα πρέπει να βάλουμε άλλα 5, να κινητοποιήσουμε άλλα 5 δισεκατομμύρια σε πραγματικά χρήματα για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα της ε, εγγύησης. Είναι σωστή αυτή η, αυτός ο υπολογισμός μου, από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Δεύτερον, όσον αφορά την υλοποίηση του Ταμείου Συνοχής, ε, όπως είπε ο Πρόεδρος, Χθες ασχοληθήκαμε με τον διορθωτικό προϋπολογισμό και είδαμε αρκετά ανησυχητικά στοιχεία γιατί είδαμε την κατάσταση ε, ε, της συνοχής και μια μείωση 7 δισεκατομμύρια ε, το περασμένο έτος. Οι εξηγήσει της Επιτροπής ήταν ότι δεν μας είχαν δώσει σωστά στοιχεία τα κράτη-μέλη. Τώρα μας λέτε ε, αυξάνουμε τα χορηγούμενα κονδύλια κατά 25%. Ε, ε, αν μπορέσουν να εκταμιευθούν τόσα χρήματα, καλό είναι. Η Επιτροπή μας λέει ότι εμείς διδασκόμαστε από τα στοιχεία τα οποία μας δίνουν τα κράτη-μέλη. Εγώ το μεταφράζω αυτό σαν να μας δείτε ότι αυτά που σας λένε τα κράτη-μέλη δεν τα παίρνετε 100% της μετρητής. Μαντεύεται λίγο δηλαδή τι πρόκειται να γίνει ή κάνω λάθος. Και τελευταία παρατήρηση, 5% μείωση προσωπικού. Και κάποια στοιχεία θα προκύψουν το 2019. Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω το 2018 θα κάνουν αυτή τη μείωση. Ε, σωστά το αντιλαμβάνομαι. Ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε κλείσει με τα σχόλια. Θα επανέλθουμε ε, σήμερα. Βεβαίως έχουμε περιορισμό χρόνου ε, και μερικές απογοητεύσεις, αλλά έχετε λάβει, αγαπητοί συνέδελφοι, στα mail σας το σχέδιο προϋπολογισμού που μόλις υιοθετήθηκε από την Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, έχετε τώρα το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που τέθηκαν και να μας δώσετε τις τελευταίες σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έγιναν κάποιες σημαντικές ερωτήσεις, θέλω να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Όσον αφορά την προστασία του κλίματος, Ο δεύτερο, η δεύτερη χώρα σε σημασία εκπομπών είναι η Ευρωπαϊκή, είναι ε, οι, Ηνωμένε Πολιτείε. Οι στόχοι που συμφωνήθηκαν για το 2030 και το 2050 στο Μαρακές παραμένουν σε ισχύ. Εάν η Ουάσιγκτον αποφασίζει κάτι διαφορετικό. Σημαντικό είναι να παραμείνουμε εμείς πιστοί στους στόχους μας. Ε, διότι ε, κάποιες φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι αν εκείνοι πουν όχι, θα πούμε και εμείς όχι. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα τέτοιο στόχο, να πούμε ότι εμείς δεσμευόμαστε όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Είμαστε πεπισμένοι ότι ε, είναι χρήσιμη αυτή η στόχη. Εάν κάποιος εταίρος μας εγκαταλείψει, εμείς τους στόχους μας συνεχίζουμε να τους θεωρούμε ενισχύει. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και για τον προϋπολογισμό, Ξέρετε ότι παρότι από τεχνικής πλευράς είναι δύσκολο να γίνει ο υπολογισμός, εμείς έχουμε ένα στόχο 20%. 20% των επενδύσεών μας και των, μας, των δαπανών μας συγγνώμη, για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία ελέγχει η Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού και το Ελεγκτικό Συνέδριο που έχει επαείοντες που εργάζονται επί του θέματος για το πώς αυτό το στόχο του 20% των δαπανών μπορούμε και να τον ελέγξουμε και να τον επαληθεύσουμε. Για το Erasmus Plus, θέλω να πω ότι είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα. Είμαι και εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους από την Επιτροπή υπεύθυνο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ούτως ώστε ε, να συνεχίσει να είναι επιτυχημένο το Erasmus Plus. Από το Erasmus Plus πήραμε μόνο αυτά τα κονδύλια τα οποία είχαν δεσμευτεί για, το ευρωπαϊκό, ε, για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντικής Εργασίας. Ε, δηλαδή, αναβαθμίζουμε τις εθελοντικές υπηρεσίες με ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με καλύτερη ποιότητα, με δραστηριότητα που θα διαρκεί περισσότερο και έχοντας κατά νου την αλληλεγγύη. Κατά τα άλλα, δεν αγγίζουμε το Erasmus Plus. Κάποια κονδύλια παίρνουμε από το Κοινωνικό Ταμείο, κάτι λιγότερο από το Γεωργικό Ταμείο και fresh money, χρήματα τα οποία διαθέτουμε για αυτό το σκοπό. Οι νέοι που διαθέτουν το χρόνο τους, που μέσα στην αιρή τους ηλικία δίνουν κάποιες εβδομάδες ή κάποιους μήνες για προγράμματα προστασίας της φύσης, ε, προγράμματα προστασίας των ειδών, προστασίας του περιβάλλοντος ή που εργάζονται με άτομα με αναπηρία ή που αφιερώνουν χρόνο για την ένταξη των προσφύγων. Θα θέλαμε να τους δώσουμε περισσότερα χρήματα από ό,τι τώρα, γιατί αυτό το οποίο κάνουν θα έχει και μια σφραγίδα ποιότητας. Είναι κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει και για την σταδιοδρομία τους, θα τους δώσει προστιθέμενη αξία για την υπόλοιπη ζωή τους. Για την γεωργία θεωρούμε ότι είναι επαρκή τα ε, κονδύλια τα οποία διατίθενται. Λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι βάσει της ε, πείρας μας από τα προηγούμενα χρόνια. Και ο υπολογισμός μας γίνεται με προοπτικές τις οποίες έχουμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι παραμένουμε απόλυτα ρεαλιστικοί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το πρόγραμμα COSME το 2017 είχαμε εξαιρετικά υψηλές δαπάνες. Το 2018 δεν κάνουμε περικοπές, απλώς επιστρέφουμε στην δομή η οποία ήταν ούτως ή άλλως η αναμενόμενη. Το 5% μείωση διοικητικών δαπανών είχε συμφωνηθεί ότι θα γίνει μέχρι τα τέλη του 2017. Και η Επιτροπή τήρησε αυτό το στόχο και κάνει τις περικοπές μέχρι το τέλος του 2017. Ορισμένα θεσμικά όργανα, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποιοι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την Επιτροπή συμφώνησαν να γίνουν αυτές οι περικοπές μέχρι το τέλος του 2018. Είναι μια ευελιξία η οποία δεν δημιουργεί νομίζω ανησυχίες. Επιστρέφω τώρα στο θέμα των πιστώσεων πληρωμών. Ε, βασιζόμαστε στις πληρωμές ε, οι οποίες γίνονται από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες, ε, οι κοινότητες, οι τοπικές αρχές και διοικήσεις Τα προγράμματά μας δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τα κράτη-μέλη. Η κοινή γεωργική πολιτική έχει αποφασιστεί στο Συμβούλιο, είναι η κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά υλοποιείται από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις που είναι πιο κοντά στους αγρότες, κοντά στους πολίτες. Και όταν μιλάμε για το greening, αυτοί θα το ελέγξουν επί τόπου, αυτοί θα λειτουργούν τα προγράμματα. Κάθε κράτος μέλος γνωρίζει τι του αντιστοιχεί κάθε χρόνο. το πρόγραμμα συνοχής και τα διάφορα προγράμματα αποφασίστηκαν στο τέλος του 2013, πολύ καθυστερημένα δηλαδή. Θα ήθελα να μπορέσουμε να αποφασίσουμε το ε, επόμενο πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο με εσάς, το Κοινοβούλιο. Εκεί να συμφωνείτε κι εσείς και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή Μπαρόζο είχε καταθέσει τις προτάσεις τον Ιούνιο του 2011 και ο κύριος Λεβαντόφσκι ε, πριν από μένα. Αλλά ήταν χαμένος χρόνος αυτός που πέρασε μέχρι το τέλος του 2013. Δύο χρόνια αργότερα μπόρεσε να γίνει σωστά αυτή η συζήτηση. Αυτό είναι κακή δημοσιονομική διαχείριση, είναι κακή διακυβέρνηση, δεν είναι χρηστή διακυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν μαζί, γιατί εγώ θα ήθελα με αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου να μπορέσουμε να το συζητήσουμε, να το λάβουμε υπόψη μας αυτό που έγινε την προηγούμενη φορά και να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις επόμενες, το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το συντομότερο δυνατόν και να λάβουμε υπόψη και τις συνέπειες του Brexit και του χρόνου το καλοκαίρι Σημειώστε το αυτό, πείτε το στους αρμόδιους συναδέλφους σας. Το καλοκαίρι του χρόνου θα πρέπει να μπορέσουμε να συζητήσουμε το επόμενο πολίτες, δημοσιονομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένο των συνθηκών του Brexit εμείς είμαστε ανοιχτοί ως Επιτροπή. Η χρηστή διακυβέρνηση απαιτεί να μην έχουμε τέτοια καθυστέρηση όπως είχαμε από το 2011 μέχρι το 2013. Εμείς ελέγχουμε τα προγράμματα, τα έργα που συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα. Ελέγχουμε πιθανές, πιθανά ενδεχόμενα ε, κακοδιαχείρισης. Αλλά όταν φτάσουμε στο θέμα της εξόφλησης των δαπανών, είναι και τα κράτη-μέλη εμπλεκόμενα μέρη. Η αύξηση την οποία δίνουμε εμείς σε αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού θεωρώ ότι είναι ρεαλιστική, διότι έχουμε φτάσει τώρα στην ταχύτητα στην οποία τρέχουν τα προγράμματα. Πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη διαχειρίζονται τα προγράμματα. Στην πρόταση που υποβάλλουμε βλέπετε τις αυξήσεις που, που έχουμε προτείνει για τα διάφορα προγράμματα και για το Εράσμους και για το Ορίζον, προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία εσείς μας είχατε εκφράσει ως προσδοκίες εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι προβλέψατε να έρθετε τις 28 Ιουνίου στην Επιτροπή Προπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μιλήσετε πάνω σε ένα έγγραφο προβληματισμού που θα αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ο προϋπολογισμός είναι ο καθρέφτης των επιλογών της Ένωσης. Θα έρθετε επίσης και στις 20 Ιουνίου για να μιλήσετε για το επόμενο πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο στις, φυσικά στις 28, όπως μόλις είπα. Φυσικά το μήνυμά σας ε, έχει περάσει για, το πρόγραμμα, για τα προγράμματα. Όταν έχουμε το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και όταν καθορίζονται τα νέα προγράμματα από την ε, Κομισιόν και το Συμβούλιο, χρειάζονται πάντα χρόνος, ούτως όντι τα κράτη, οι δήμοι, οι κοινότητες, να αισθανθούν ότι είναι δικά τους τα προγράμματα και να τα εγκολποθούν, ας πούμε, και χρειάζονται δύο-τρία χρόνια γι' αυτό. Τώρα, έφτασε η ώρα να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε τόσο γρήγορα μετά την ε, ειδοποίησή μας, γιατί σήμερα το πρωί μόλις ε, μίλησε για αυτό το θέμα ε, το Σώμα των Επιτρόπων και ενέκρινε το σχέδιο προπολογισμού για τον προπολογισμό του 2018. Και αν δεν έχετε άλλε παρατηρήσει, λύεται εδώ η συνεδρίαση. Θα συνεδριάσουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη 19 και 20 Ιουνίου και θα κάνουμε μια έκτακτη συνεδρίαση στις 28 Ιουνίου μόνο το απόγευμα. Τελειώνει εδώ η συνεδρίασή μας.